συζητήσεις για αλλαγή και διορισμό σε επιτροπές. Αυτές ε, τις, ε, τους διορισμούς θα τους ε, δημοσιεύσουμε στα πρακτικά και αν δεν υπάρχουν στάσεις στους διορισμούς αυτούς